των κυρίων Σοσνιέρ και Γκάμπελιτς που ε, λαμβάνουν έναρξη 22 Μαρτίου 2018 και 4 Απριλίου 2018 προς αντικατάσταση των κυρίων Κόρβιν Μίκε και Νίλσον. Ε, καλωσορίζω τους συναδέλφους και θυμίζω ότι αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους πλήρως στο Κοινοβούλιο βάσει των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τον ιστορικό κανονισμό. Μετά τις εκλογές των κυρίων ε, Τζάνι Πιτέλα και Ματέο Σαλβίνη ως γερουσιαστών της Ιταλικής Δημοκρατίας και του κυρίου Λορέντζο Φοντάνα στην Εθνική Βουλή τη Ιταλία, το Κοινοβούλιο βάνει γνώση ότι οι θέσει του χειρεύουν από τι 23 Μαρτίου 2018. Μετά την παρέτηση του κ. Ζανπόλ Ντενανό, το Κοινοβούλιο βάσει του κανονισμού ε, από την χειρία τη ε, θέση του από τι 11 Ιουνίου 2018 θα ενημερώσει τι αρμόδιε εθνικέ αρχέ.